του κανονισμού μας στις αρμόδιες αρχές και θα δημοσιευθεί στα σχετικό έντυπο. Η γραπτή δήλωση των ε, κυρίων Φιώνα Χόλι, Νέσα Γελασέντερ, Ιζαμπέλ Τουγόν, Δίτερ Λέμπρεχτ Κόχ και Σαμπίν Βίλς ως προς τα ατυχήματα βαρέων οχημάτων έχει συλλέξει τις υπογραφές ε, της πλειοψηφίας και άνω των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού μας ε, θα διαβιβαστεί σε αρμόδιες αρχές και θα δημοσιευθεί στα υιοθετηθέντα κείμενα. Και τώρα ο κύριος Νάτρας έχει στήσει το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ με αυτά που έχουμε συζητήσει, θα θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ασφάλεια μας στα κτίρια μα Θα ήθελα να απευθύνω και εγώ ευχαριστήσω προς το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά μα και θέλω να ζητήσω να διερευνηθούν ε, περιπτώσεις παραβίασης ασφάλειας των όρων ασφαλεία τη Βρυξέλλες και κυρίω τη χρήση, κατοχής και χρήσης ε, πυροβόλων όπλων. Έχουν διερευνηθεί τα πράγματα γιατί πρόκειται για ζητήματα τα οποία θέτουν την προσωπική μα ασφάλεια, αλλά την ασφάλεια και του προσωπικού και των επισκεπτών μα σε κίνδυνο θα πρέπει να ε, ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, αλλά ελπίζω να μην, ε, τεθούν, να μην θυσιαστούν οι στρατιώτες προκειμένου να διαφυλαχθεί η θέση και ο φόκος ορισμένων στρατηγών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία συνεχίζεται ε, αδιάλειπτα για να ενισχυθεί η ασφάλεια στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Ταραμπέλα, 720. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα στο πλαίσιο της ε, υπογραφής ε, της δήλωσης 84 να ευχαριστώ τους αδέλφους Μπαστός, Κανφά, Βερσιά, Βέμπερ από τους Πρασίνους, τους ε, το έλκα ε, για τις υπογραφές τους και να ευχαριστώ και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν για την αποστολή αυτού του σοφούς μηνύματος ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ζητούμε ένα κοινό καταστατικό για τις αλληλασφαλιστικές εταιρείε, τους συνεταιρισμούς και τα ιδρύματα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Προχωρώ τώρα στις ψηφοφορίες. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την, πρόταση, την ψηφοφορία για δύο προτάσεις ψηφίσματος για τον Ουγγρικό νόμο για τη Μέσα Ενημέρωση. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν την ψηφοφορία που προβλέπετε για το ψήφισμα για τα ΜΜΕ στην Ουγγαρία, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή